Περάσουμε στην πρώτη ψηφοφορία, έκθεση Stevens, με ονομαστική κλίση. Μία ενιαία ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία, παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνατε και σας ευχαριστώ. Περνάμε στη δεύτερη έκθεση, έκθεση Μπόνι. Με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται. Τρίτη έκθεση της κυρίας Χιμένας Μπεσερίλ με ονομαστική κλίση και πάλι. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Δεύτερη έκθεση της κυρίας Μπεσερίλ με ονομαστική ψηφοφορία, έρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, τέλος. Εγκρίνεται. Δεύτερη έκθεση τώρα του κυρίου Μπόνι, με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Έκθεση Νοβάκοφ. Με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Έκθεση Ροζιέρ. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχιτη ψηφοφορία. Αν ψηφίσατε όλοι, ε, Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η έκθεση Ροζιέρ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Ροζιέρ για να μας πει δύο λόγια μετά το πέρας ψηφοφορίας της έκθεσής της. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που συνέβαλαν στην υπερψήφιση της έκθεσης ε, για την αγαστή συνεργασία που είχαμε και το πολύ καλό κλίμα τους τελευταίους μήνες και εβδομάδες. Και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει συνέχεια στην έκθεση προτείνοντας νομοθετική πρόταση όπως απευθύναμε και έκκληση στην έκθεσή μας. Ωραία, ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στην έκθεση Μιχαήλωβα. Ψηφίζουμε τροπολογία 8. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9 της κυρίας Μιχαήλοβα, ε, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 10, ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 11 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 3, ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 1, με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ε, συγγνώμη, ξέχασα να ρωτάω για αποχές. Τροπολογία 2 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα με ονομαστική κλίση το νομοθετικό ψήφισμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ. Περνάμε στην έκθεση Γκάιερ με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Ρούμπιχ. Μία ψηφοφορία, ονομαστικά άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και η έκθεση Ρούμπιχ. Περνάμε στην επόμενη που είναι τη κυρία Βάνα. Με ονομαστική κλίση μια ενιαία ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και επόμενη έκθεση κυρία Θεοχάρους. Παράγραφος 28 σε δύο τμήματα. Ψηφίσουμε το πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Για το δεύτερο τμήμα της παραγράφου 28 άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται όντως. Ψηφίζουμε το ψήφισμα τώρα. Ονομαστικά έρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες.